Hello, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Αν μπορείτε να καθίσετε όλοι. Το πρώτο στοιχείο της ημέρας διάταξής μας είναι η έγκριση της ίδιας ημέρας διάταξης. Αν δεν έχετε καμία αντίληση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η ημέρας διάταξη και στη συνέχεια είναι η ανακοινώση Προέδρου. Καθόλου δεν έχω να σας ανακοινώσω τέτοιες ανακοινώσεις. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 και 29 Σεπτεμβρίου ενεστώτος. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε σχέση με τα πρακτικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Τέταρτο σημείο της σημερινής διάταξης είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γιάνν Ντεβίτ, πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας για το Χρηματοοικονομικό Σύστημα από την Ανοβουλή του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μπορώ να, παρα... να παρουσιάσω στην Επιτροπή μας τον κύριο Ντεβίτ, ο οποίος έχει κάνει νομικές σπουδές, υπήρξε δικηγόρο στην... στις κάτω χώρες πρωτού, γίνει μπει στην πολιτική ζωή στο Συμβούλιο του Χέρλεν, μετά έγινε βουλευτή το 1995 και στην κάτω και στην Ανοβουλή και από το 2009 είναι πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας για το Χρηματοοικονομικό Σύστημα της Δεύτερης Βουλής της Άνω δηλαδή του Κοινοβουλίου των Κάτω Χωρών. Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ εδώ, εξ ονόματος του Πρόεδρου μας, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα. Η Επιτροπή σας δημιουργήθηκε στην ε, Ολλανδία τον Ιούλιο του 2009 και έχει εκπληρώσει το πρώτο τμήμα του έργου της που ήταν η έρευνα στις έρευνες του, της χρηματοοικονομικής κρίσης, των διαφορετικών προβλημάτων και των μέτρων που ελήφθησαν στις κάτω χώρες. Το πρώτο τμήμα της έκθεσης έγινε δεκτό από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο του Σεπτέμβριο και τώρα η Επιτροπή έχει περάσει στη δεύτερη φάση του έργου της, που είναι μια έρευνα της παρέμβασης της Ολλανδικής Κυβέρνησης ε, στις χρηματαγορές από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι σήμερα. Σας δίνω λοιπόν με μεγάλη χαρά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής ε, για την χρηματοοικονομική κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνεται είναι μεγάλη χαρά για μένα να μπορέσω να παρουσιάσω την έκθεση της Επιτροπής μας στη Δεύτερη Βουλή των Κάτω Χωρών και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήματα που θα έχετε. Θέλω να σας παρουσιάσω μια σειρά από διαφάνειες και να σας εξηγήσω ποια ήταν τα πορίσματα της έρευνάς μας. Πρωτού όμως περάσουμε σε αυτό το στάδιο, Θέλω να σας παρουσιάσω τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται μαζί μου, Γιώργ Τάμερ στα αριστερά μου και Χέρμαν Μπέρν και οι δύο ερευνητέ. και στο βάθος της αίθουσας Χέν Βαντελάιτε και Λαταλή Κότ που ήταν η συντονίστρια αυτή, ήταν οι συντονιστές μάλλον δυο τους της έρευνας αυτής. Και επίσης, πρωτού συνεχίσω κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα εξώματος του Ολλανδικού Κοινοβουλίου να σας δώσω ένα πρωτότυπο αντίγραφο αυτής της έκθεσης μαζί με τα ε, παρατήματά του. Δυστυχώς είναι στα Ολλανδικά και μάλλον θα το θέσετε στην βιβλιοθήκη σας χωρίς περαιτέρω ανάγνωση. Είναι και βαρύ κιόλας το, το ευλογημένο αυτό έγγραφο. Ωραία. Τούτου λεχθέντος και πραχθέντος θα ήθελα σας προτείνω να κάνουμε μια επισκόπηση των ε, αποτελεσμάτων της ερευνάς μας και των συστάσεων που έχουμε εκδώσει μετά από την έρευνα αυτή. Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθώ στην σύνθεση και τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρός σας πριν από λίγο, θα ήθελα να εξηγήσω καταρχήν τον τρόπο λειτουργία μα. δύο, υπάρχουν δύο τμήματα αυτής της έρευνας. Το πρώτο τμήμα αφορούσε την ανατομή των αιτιών της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως στον τομέα της στον πιστοτικό τομέα, ενώ στο δεύτερο τμήμα της έρευνας θα ασχοληθούμε με τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει, τι έγινε και τι πρέπει να γίνει με τα εκατομμύρια που έδωσε η χώρα μα στις τράπεζες και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Οκτώ κοινοβουλευτικοί ήταν στην Επιτροπή μα, εκπροσωπώντα οκτώ πολιτικά κόμματα που είναι παρόντε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Τότε βέβαια υπήρχαν 11 κόμματα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, μόνο οκτώ από τα οποία ήταν παρόντα στην ε, ερευνητική μας επιτροπή. Εμείς, όπως είπε και η πρόεδρο. Έχουμε <clears throat> ξεκινήσει τις εργασίες μας τον Ιούλιο του 2009 με την εντολή να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της ε, ε καταιγίδα ουσιαστικά που έλαβε χώρα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από το 2009 και επίσης τμήμα της ε, εντολής μας ήταν το να διατυπώσουμε προτάσεις για τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να μην υπάρξει και επανάληψη αυτού του δράματος που ζήσαμε όλοι τα δύο τελευταία χρόνια. Η έρευνά μας ε, έχει δύο τμήματα, όπως είπαμε. Σήμερα θέλω να αναφερθώ κυρίως στις αιτίες της κρίσης και στα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει εμείς. η έκθεσή μας. Εν έχει συζητηθεί από, το, από την δεύτερη Βουλή του Ουρανικού Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο και οι συστάσεις της ενεκρίθησαν ομοφόνος από την Βουλή αυτή. Ποιες είναι λοιπόν οι αιτίες της κρίσης αυτής. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η κρίση έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Είναι μια κρίση η οποία είχε και την ευρωπαϊκή της διάσταση και εδώ θέλω να εστιάσω ιδιαίτερα στην κατάσταση που αντιμετωπίσαμε στις κάτω χώρες. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια ήταν η θέση του νομοθέτη, των νομοθετικών αρχών στην ε, Ολλανδία και των εποπτικών αρχών για τις αγορές. Και φυσικά η έρευνά μας εξετάζει συγκεκριμένα την κατάσταση στη δική μας χώρα. Για να μπορέσουμε να προβούμε σε κάποια ανάλυση αυτών των αιτίων, μελετήσαμε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, πάντα τη αιτήση της Δεύτερης Βουλής, την ε, εξαγορά του ομίλου ABN AMRO από το ε, Consortium Fortis Τράπεζα του Σαντανδέρ Όπως ξέρετε αυτή η διαδικασία έλαβε χώρα το 2007 και μετά είχαμε επίσης και την κατάρρευση της ε, Ισλανδικής Τράπεζας και της iSave η οποία κατέρευσε το 2008 οδηγώντας σε πολλά προβλήματα στις κάτω Στη δεύτερη αυτή συγκεκριμένη περίπτωση θέλησαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των δημοσίων αρχών στι κάτω χώρε. Δηλαδή πώ λειτουργήσε το Υπουργείο Οικονομικών και Εθνική Οικονομία στι κάτω χώρε και ποιο ήταν ο ρόλο του τραπεζικού συστήματο στι κάτω χώρε και των αρχών ρυθμιστικών για την αγορά. Αλλά όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει κυρίως ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος και του Ολλανδού Υπουργού Οικονομικών. Ε, μέθοδος εργασίας τώρα. Καταρχήν, με το προσωπικό μας και τους συνεργάτες μας κάναμε μία μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, διότι πράγματι έχουν συγγραφεί πολλά βιβλία και πολλά άρθρα σε σχέση με την κρίση αυτή την οικονομική και χρηματοοικονομική και κάναμε επίσης και μια σειρά από συνεντεύξεις με προσωπικότητες, με εμπειρογνώμονες με άτομα τα οποία έχουν προεξάρχοντα ρόλο στον οικονομικό στίβο και τα οποία γνωρίζουν πολύ, πολύ καλά την κατάσταση. Επίσης, πολλές από τις ε, ακροάσεις μας έγιναν με ε, ζωντανή, μεταδόθηκαν ζωντανά από το πρώτο Ολλανδικό κανάλι τηλεόρασης. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες και ε, δυνατές πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών και από τις διάφορες τράπεζες με τις οποίες είχαμε σε επαφή. Και φυσικά δημιουργήσαμε και μία δεξαμενή σκέψη κατά κάποιο τρόπο, μία αν θέλετε συμβουλευτική ομάδα με την ε, αρρωγή του Πανεπιστήμιου του Άμστερνταμ, του Πανεπιστήμιου του Τίλμπερκ, και επίσης με την αρρωγή ενός διευθυντή ε, Ταμείου Συντάξεων στις κάτω χώρες. Ποια είναι τα συμπεράσματά μας. Είδαμε καταρχήν ότι η παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική, κρίση καλύτερα είχε σχετικά σαφή αίτια. Όλα τα μονοπάτια έρευνας μας οδηγούν στην στεγαστική αγορά των ΗΠΑ. Έλαβε χώρα μια τεράστια έκρηξη αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ, συγχρόνως όμως και μια τεράστια αύξηση και πολλαπλασιασμός του αριθμού των στεγαστικών υποθηκών. Μαζί με τις διαταραχές της αγοράς, όλα αυτά οδήγησαν σε μια, σε μια φυσαλίδα χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τώρα τις μακροοικονομικές αιτίε, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες ήταν οι εμπορικές και νομισματικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν το διάστημα πριν από την κρίση. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν χώρα σημαντικές ε, εισαγωγές, υπήρξε μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συλλαγών στι ΗΠΑ και αντίστοιχα μεγάλο, μεγάλο πλεόνασμα από τη μεριά τη Κίνα. Όλα αυτά οδήγησαν σε αυξανόμενο δανεισμό στι ΗΠΑ με τα συμπεράσματα αυτά που έχουμε. Επίση, υπήρξε αυξανόμενη απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών ε, αγορών και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη με αποτέλεσμα οι χρηματαγορέ να έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία δράσης και οι συνέπειες αυτής της ε, απελευθέρωσης ήταν χαμηλά επιτόκια, μεγάλη οικονομική μεγέθυνση, μεγάλη αύξηση της ε, δανειοδότησης με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Υπήρξαν λοιπόν υψηλοί κίνδυνοι τους οποίους ανέλαβαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μας οδήγησαν στην κατάρρευση που γνωρίζουμε όλοι. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμά μας, η καλύτερη υπότιση σύσταση που έχουμε απευθύνει προς την κυβέρνηση των κάτω χωρών, είναι ότι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα από τα αίτια της κρίσης η έλλειψη προβλέψεων. Κανείς δεν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να διακρίνει τα ίχνη της επερχόμενης κρίσης. Μία φορά το χρόνο ζητήσαμε επομένω η Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών και το Γενικό Γραφείο Σχεδιασμού να κάνουν μια έκθεση σε ετήσιο επίπεδο όπου θα γίνεται ένας απολογισμός της κατάστασης των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χώρα μας. Η χώρα αυτή λοιπόν δεν θα πρέπει να αναφέρεται μονάχα στι μακροοικονομικέ παραμέτρου και την κατάσταση αυτή στη χώρα μα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζει γενικότερα την κατάσταση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματο τη χώρα μα εν γέννη. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να απευθύνεται στο Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών. Και ο στόχο τη θα πρέπει να είναι να εξηγεί ποια είναι η κατάσταση στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ και ποια είναι η μακροοικονομική κατάσταση. Επίση, Θέλησαμε να αναλύσουμε ποιοι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι συνέτειναν στην κρίση. Καταρχήν, οι τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήταν ότι οι τράπεζες αποδίθηκαν σε ενέργειες οι οποίες ήταν επικίνδυνες ακόμα και τυχοδιοκτικές. Υπήρξε υποτίμηση του κινδύνου και οι κίνδυνοι αυτοί πολλές φορές ανελήφθησαν εν γνώση του επίπεδου κινδύνου. Υπήρξε μια προσπάθεια λοιπόν να ε, καταμετρηθεί το επίπεδο κινδύνου, αλλά υπερκέρασαν την εκτίμηση του κινδύνου πολλές φορές οι, τα συμφέροντα, τα εμπορικά και τα οικονομικά των τραπεζών. Ένα άλλο στοιχείο ήταν η ολοένα αυξανόμενη πίεση των μετόχων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τραπεζών. Οι μέτοχοι θέλουν να υπάρξει δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μία αύξηση επομένως του, της αξίας των μετοχών τους. Αυτό οδήγησε σε στρεβλωτικά αποτελέσματα στις τράπεζες. Συγκεκριμένα έγιναν πολύ πιο σημαντικά τα πριμ, τα μπόνους που έπαιρναν τα στελέχη των τραπεζών από ότι έπαιξαν πιο μεγάλο ρόλο στην συμπεριφορά λοιπόν των στελεχών των τραπεζών τα μπόνους από ότι η σωστή εκτίμηση του κινδύνου. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος και η εκτίμηση κινδύνου στις τράπεζες είχαν ένα χαρακτήρα στρεβλό. Τα συμβούλια και οι διάφοροι φορείς εκτίμηση του κινδύνου δεν έπαιξαν τον απαραίτητο ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να επανεξετάσουμε το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης των ε, ελεγκτικών, των εσωτερικών ελεγκτικών αρχών μέσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει λοιπόν σε μια αναθεώρηση των ε, ρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Γνωρίζετε ότι υπάρχει και ένας τραπεζικός κώδικας στις κάτω χώρες, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά από την ε, κρίση και ο οποίος έχει σαν στόχο να καθορίζει τους κανόνες στο εσωτερικό των τραπεζών. Περιλαμβάνει λοιπόν ο κώδικας αυτός ε, κανόνες για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των εσωτερικών ελεγκτών σε κάθε πιστοτικό ίδρυμα. Περιλαμβάνει λοιπόν και μνήες και αναφορές στην ε, αμοιβή των τραπεζικών στελεχών. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε μέσα σε αυτό τον κώδικα είναι ότι αφεαυτό ο κώδικας αυτός δεν επήρκεσε. Η διαχείριση του κινδύνου από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στον κώδικα αυτό. Επίσης, η αμοιβή των ανωτέρων στελεχών δεν καθορίζεται παρά μόνο στο υψηλότερο επίπεδο της τραπεζικής ιεραρχίας. Θεωρήσαμε ότι τα πριν και οι αμοιβέ των στελεχών θα πρέπει να την χάνουν ρύθμιση για το σύνολο των στελεχών του οργανογράμματος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επομένως θεωρήσαμε πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω αυτός ο τραπεζικός κώδικος, κώδικς και να συνδεθούν οι προβλέψεις του και οι πρόνοιές του με συγκεκριμένες κυρώσεις, εάν οι τράπεζες δεν ακολουθούν και δεν σέβονται αυτό τον κώδικα. Και τώρα, μετά από νομοθετικές ρυθμίσεις του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, γιατί έχει ξεπεραστεί πια η φάση της αυτορύθμισης, υπάρχει μια σειρά από μέτρων τα οποία διέπουν τη λειτουργία των τραπεζών και επίσης ορίζουν το επίπεδο των αμοιβών και των πόνους των στελεχών. Και ζητήσαμε να υπάρξει και μεγαλύτερη ισχύς και δυνατότητα δράσης των εσωτερικών έλεγχων ε, ελεγκτών, γιατί διαπιστώσαμε ότι σε πολλές φορές οι εσωτερικοί αυτοί οι ελεγκτές δεν είχαν πολύ καλή ιδέα του ρόλου που είχαν ως επόπτες και ως υπεύθυνοι για να κρούσουν τον κώδικα του κίνδυνου. Θεωρούμε επίσης ότι και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός των τραπεζών θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα αντίστοιχο κώδικα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή τα συνταξιδοτικά ταμεία κτλ. Νομίζουμε ότι ο κώδικας αυτός θα πρέπει να έχει ένα ανάλογο χαρακτήρα και για του φορεί αυτού όπω είναι οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Επίση, αντιμετώπισαμε και το ρόλο των νομοθετικών αρχών μέσα στα πλαίσια τη κρίση αυτή, τη πιστοτική. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι οι ρυθμίσει οι οποίε εφαρμόστηκαν στι κατοχώρε είχαν σαν κύριο στόχο την εναρμόνιση και την απελευθέρωση το, της χρηματοπιστωτικής αγοράς της κάτω χώρες, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να βρίσκεται σε ίσο επίπεδο ανταγωνισμού με άλλες διεθνείς αγορές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι λησμόνισαν ορισμένα ασθενή στοιχεία του συστήματος οι ρυθμιστές και νομοθέτες. Παραδείγματος χάρη τις κεφαλουχικές απαιτήσει οι οποίες είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ορισμένες τράπεζες πήρανε αλόγιστους κινδύνους, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και διαπιστώσαμε επίσης ότι οι λογιστικοί κανόνες λειτουργούν με υπερκυκλικό τρόπο. Και αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της κρίσης. Γι' αυτό έχουμε προτείνει μια σειρά από μέτρα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Εξάλλου, εκτός του τραπεζικού και πιστοτικού συστήματος που υπόκειται σε ρύθμιση, υπάρχει ο λεγόμενος σκιώδης τραπεζικός τομέας. Ο υπόγειος τραπεζικός τομέας που δεν υπόκειται σε ρύθμιση. Δηλαδή είναι φορείς και ιδρύματα τα οποία δεν είναι τράπεζες αλλά παίζουν ένα ρόλο στο ε, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν δεν είχε μια ιδιαίτερα κριτική στάση απέναντι σε εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο θεωρήσαμε ότι η φιλελευθερωποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών δεν έτυχε επαρκούς ελέγχου και κανείς δεν σκέφτηκε προς τα πού μας πηγαίνει αυτή η πορεία φιλελευθερωποίησης. Επίσης, θεωρούμε ότι δεν υπήρξε παρακολούθηση της εξέλιξης κατάστασης από τις νομοθετικές αρχές. Πολλές φορές το Κοινοβούλιο μας έπαιξε το ρόλο ενός παθητικού παρατηρητή, ο οποίος δεν ελάμβανε χώρα της εξελίξη κινήσεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη παρεμβατικότητα από την πλευρά του. Έχουμε υποβάλει και μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις εξάλλου. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ω εκ τούτου, η επίλυση του προβλήματος και οι ρυθμίσει θα πρέπει να γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει επαρκώ σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον θα πρέπει να το πράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν δεν μπορεί να προχωρήσει επαρκώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την επανάληψη τη κρίση που γνωρίσαμε. Δεύτερον, προτείνουμε μία αύξηση του λόγου ε, και επομένως μια αύξηση του ιδίου κεφαλαίου των τραπεζών. Επομένως, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να υπάρξει εφαρμογή των κανόνων που έχει προτείνει η Επιτροπή τη Βασιλείας. Προτείνουμε επίσης να υπάρξει μέσα στις ίδιες τις τράπεζε μία, ένας διαχωρισμός των ενεργειών κλασικής τραπεζικής λειτουργίας από τις δράσεις οι οποίες έχουν χαρακτήρα ε, χρηματοοικο... Ε, λειτουργίας της χρηματαγορές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν οι καταθέσεις των ε, απλών καταθετών να εμπλέκονται σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Να υπάρχει λοιπόν μια απόλυτα χωριστή λειτουργία της τράπεζας καταθέσεων, του τμήματος της τράπεζας που έχει να κάνει με τις καταθέσεις των απλών καταθετών, από τις ενέργειες της χρηματαγορές, ώστε να μην είναι οι καταθέτες αυτοί οι οποίοι θα πληρώνουν την ύφη για τις απώλειες της χρηματαγορές. Και έρχομαι τώρα σε έναν χώρο, ο οποίος ίσως είναι πολύ πιο γνωστός σε εσά. Είναι η οδηγία Αντών Βενετά. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα αυτήν την ε, οδηγία σε επίπεδο κοινοβουλίου. Αλλά η οδηγία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά κριτηρίων σε περίπτωση εξαγοράς, συγχώνευσης τραπεζικών ε, Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν επανεξέταση της σταθερότητας και της φερεγγιότητας ενός φορέα μετά από μια ενέργεια εξαγοράς ή συγχώνευσης. Έλεγα λοιπόν για την περίπτωση της ε, εξαγοράς της Αμορα από, από τον Πάνκο Σαντανδέρ και την Fortis είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει εκ νέου επαλήθευση της ασφάλειας και της συστημικής ευρωστίας μιας τράπεζας μέσα στα πλαίσια της οδηγίας Αντών Βένετα για να αντιμετωπίζονται προβλήματα τα οποία μπορούν να απορρέουν από συγχωνεύσεις εξαγορές επιχειρήσεων. Επίσης, και αναφέρομαι πάλι στην Ολλανδική ε, πραγματικότητα, είχαμε προτείνει η Κεντρική Τράπεζα να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης και εποπτείας στο σύστημα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από μέτρα παρέμβασης τα οποία θέλουμε να προτείνουμε τα οποία ποικίλουν από μία απλή υπενθύμηση, όχληση, προειδοποίηση προς τις τράπεζες μέχρι μέτρων τα οποία μπορεί να είναι απόλυτα δεσμευτικά όπως η εθνικοποίηση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις των καταθέσεων επίσης. Προτείνουμε να ακολουθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένα. Να υπάρχουν ε, συμβολές των ε, χρηματοπιστωτικών ε, φορέων που θα καταβάλουν εξ άντε, εκ των προτέρων, συνεισφορές στο Ταμείο Αυτό που να βασίζονται στην εκτίμηση του κινδύνου και θεωρούμε ότι πρέπει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο μετά από τις επικρίσεις που έχουμε διατυπώσει να αναλάβει την συνέπεια των πράξεών του και να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο για την προστασία από τις κρίσεις. Προτείνουμε λοιπόν το Ολλανδικό Κοινοβούλιο σε τακτικό επίπεδο και περιοδικά να εξετάζει την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να μην καταλαμβάνεται εξαπίνης όπως το παρελθόν και επομένως να μην έχει να αντιμετωπίσει οξύε κριτικές όπως αυτές που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τώρα. Εγώ θα συνεχίσω όσο θέλετε, κυρία Πρόεδρε. Αν θέλετε να με σταματήσετε, με σταματάτε. Συνεχίζω λοιπόν. Για το ρόλο των εποπτικών αρχών και των άλλων πρωταγωνιστών. Ε, Στην Ολλανδία είναι η Τράπεζα της Ολλανδίας. Η Τράπεζα της Ολλανδίας ως υπόπτες δεν απέδωσε αρκετή προσοχή στους συστημικούς κινδύνους. Έκανε μια προειδοποίηση, αλλά τίποτε παραπάνω. Δεν πήρε μέτρα. Δεν απέδωσε τη δέωσα προσοχή στους πραγματικούς συστημικούς κινδύνους. Οι επόπτες αναφέρθηκαν στην προσοχή του στην μικροεπιτήρηση διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν αναγνώρισαν ότι συνέβαινε κάτι πολύ παραπάνω και ότι υπήρχε συστημικός κίνδυνος. Επίσης διαπιστώσαμε ότι λόγω των απαιτήσεων απορρίτου μεταξύ της τράπεζας της ε, Λανδίας και των επιμέρους τραπεζών η Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο δεν είχε σαφή εικόνα του τι συνέβαινε σε μικρό επίπεδο. Και είχαμε ένα πρόβλημα. Θα το δείτε και αλλού αυτό. Είχαμε προσκρούμε, προσκρούμε στην ανάγκη του απόρριτου. Ιδιαίτερα στη σχέση των εποπτείας Κοιτάξαμε τις λογιστικές υπηρεσίες και διαπιστώσαμε ότι η σύνταξη λογαριασμών δεν απέδει ιδιαίτερη σημασία στη σύνταξη των ετήσιων λογαριασμών, ετήσιων εκθέσεων μάλλον, και τα διευκρινιστικά σχόλια. Δεν τα πρόσεχαν αυτά, ότι δηλαδή υπάρχουν κινδύνους, κίνδυνοι συγγνώμη, στα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι πολύ πιο επικριτικοί οι ελεγκτές έτσι ώστε οι αιτήσει εκθέσεις να παρουσιάσουν με σαφήνεια την κατάσταση κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, να δείχνουν ποια από τα στοιχεία ενεργητικού είναι πιο επισφαλή, τι κίνδυνοι υπάρχουν και προτείνουμε να φροντίσουμε να υπάρχει μία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή με εξουσίες επιβολής εκτελεστικές. Στην Ολλανδία υπήρχε ένα πρόβλημα μεταξύ των Ολλανδικών και των Ισλανδικών εποπτικών αρχών. Η Ολλανδία δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα του iSafe έγκαιρα, εν μέρη λόγω του ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές εποπτικές αρχές. Η κάθε μία είχε το δικό της συμφέρον. Το να έχουμε λοιπόν μια ενιαία Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για να φτάσουμε ως εκεί χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Στις συστάσεις από 20 και μετά μιλάμε για την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας. Στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ολλανδίας, μεταξύ της Υποπτικής Αρχής και του Διαμεσολαβητή για τι ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε. Εκεί μπορεί να ε, απευθυνθεί ο πολίτης αν έχει προβλήματα. Χρειάζονται ορισμένα εργαλεία υποπτικού χαρακτήρα η εργασία των, υποπ... των υποπτικών αρχών πρέπει να βελτιωθεί. Και αιτήθηκε θέμα ευθύνης των εποπτών. Στην Ολλανδία μερικές φορές Φαίνεται να μην υπάρχει αρκετή ισχύς στο όργανο αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι η αποπτική αρχή πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που ισχύει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή ο κίνδυνος της ευθύνης να μην αναφέρεται ως δικαιολογία για την μη λήψη μέτρων. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρούς κανόνες για την απόδοση ευθύνης, accountancy και ο λογιστικός έλεγχος να έχει μπροστά του σαφή κριτήρια εργασίας. Δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, ABN AMRO και iSafe. Προκειμένου να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των κανόνων που, ισχύει, που ίσχυαν και ισχύουν στην Ολλανδία, ποιος είναι ο ρόλος των επιμέρους αρχών, Από αυτό ξεκινήσαμε. Κοιτάξαμε τη θέση του Υπουργού Οικονομικών του Κοινοβουλίου και της Εποπτεύουσας Αρχής. Και τα πορίσματά για την ABN AMRO Σεπτέμβριος 2007 ήταν ότι με βάση το δεδομένο νομικό πλαίσιο ο υπουργό Οικονομικών έπρεπε να δώσει το OK για μια συγχώνευση με συμβολή της Τράπεζας της Ολλανδίας. Το θέμα λοιπόν συνετής διαχείρισης και υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τίθεται και διαπιστώσαμε ότι ο υπουργό Οικονομικών στήριξε την απόφαση του αποκλειστικά στην γνωμοδότηση της Τράπεζας της Ολλανδίας. Όσον αφορά τις ε, συνέπειες για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το ίδιο πράγμα και εδώ. Στηρίχθηκε στην Κεντρική Τράπεζα. Εδώ υπάρχει μια διαμάχη, υπάρχει μια σύγκρουση των κανόνων. Ο υπουργό ήδη ήταν έτοιμος να δώσει το πράσινο φως από την αρχή πριν την πράξη αυτή. Με βάση λοιπόν το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο, ο υπουργό δεν χρησιμοποίησε τα περιθώρια λιγμών που είχε για να βρει μια άλλη θέση και να πάρει διαφορετικά μέτρα. Δεν λέμε ότι η θα πρέπει να κάνει αυτό ή εκείνο. Λέμε ότι θα μπορούσε να είχε πάρει άλλα μέτρα. Θα μπορούσε να είχε δράσει διαφορετικά. Η δεύτερη περίπτωση είναι η Ice Save. Εδώ βρήκαμε ότι κύριος υπεύθυνος στην Landsbanki και η Ισλανδική Εποπτική Αρχή. Ένα από τα προβλήματα της... Ε, ένας από τα στελέχη μάλλον της Κεντρικής Τράπεζας στην Ολλανδία ήρθε στην Ακρόαση και μας είπε ότι είχε την εντύπωση ότι η Εποπτική Αρχή στην Ισλανδία παραπλανήθηκε. Δηλαδή σκόπιμα τους δόθηκε λάθος πληροφορία οι εποπτικές αρχές μπορεί να του συμβεί αυτό. Η τράπεζα της Ολλανδίας δεν ήταν σε θέση να εκπέμψει προειδοποίηση. Διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνο οι καταθέτες να τρέξουν στην τράπεζα και να δημιουργηθεί ένας μεγάλος κίνδυνος και ταραχή. Η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας είχε περιθώρια δράσης έναντι των προϊόντων της iSafe δεν έκανε αυτό που θα μπορούσε να είχε κάνει. Εμεί θεωρούμε ότι θα έπρεπε να, θα μπορούσε μάλλον να είχε θέσει ορισμένους όρους να τους προτείνει στο Lands για τα προϊόντα της iSafe. Δεν το έκανε αυτό επαρκώς και τελικά η Κεντρική Τράπεζα Ολλανδίας με στα πλαίσια της Ολλανδικής νομοθεσίας θα μπορούσε να είχε δώσει ενδείξεις στη Landsbanki Όσον αφορά την εποπτεία λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι αν η Τράπεζα της Ολλανδίας είχε πάρει διαφορετικά μέτρα, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. χωρίς να μπορούμε αυτό να το εγγυηθούμε 100% σε σχέση με τη Landsbanking. Τώρα, τμήμα 2. Μέτρα για την κρίση δις ευρώ που δόθηκαν από την κυβέρνηση σε διάφορα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή την πρόταση την έχει το, Ευρωπαϊκό, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα. Με βάση την έρευνα αυτή. Πιο ευρία έρευνα από την που κάναμε εμείς. Η κοινοβουλευτική έρευνα δίνει ένα ευρύτερο πλαίσιο από ό,τι η έρευνα που κάναμε εμείς. Έχουμε 6 ως 7 μέτρα που ελήφθησαν από τις Ολλανδικές Αρχές. Πρώτον, η εθνικοποίηση της ABN AMRO. Οι κεφαλογικές προβλέψεις για την ENZ, AEGON και SNS REAL. Το μέτρο εγγύησης των αρχών που πρόσφεραν οι αρχές 200 δις ευρώ οι τράπεζε και τα χρηματοπιστωτικά διδήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ποσό, να επεκταθεί το τρέχον σύστημα εγγύσεως καταθέσεων από 50 σε 500.000 ευρώ. Μετά οι διάφορες κρατικές εγγύησεις, ιδιαίτερα οι καταθέσεις της, για την, καταθέσεις της ISAVE Κάθε τράπεζα πλήρωσε μέχρι 100.000 ευρώ. Στον κάθε καταθέτη 1,3 δις ευρώ πλήρωσαν γι' αυτό οι Ολλανδικές αρχές. Και ακόμα συζητάμε πώς θα πάρουμε τα χρήματα αυτά πίσω από την Ιλλανδία και μια, ε, ένα μέσον backup για την ENZ. Το κράτος ένα έδωσε ένα είδος εγγύηση για ένα χαρτοφυλάκιο με λιγότερα προϊόντα ενυπόθηκων δανείων. Η Ολλανδική κυβέρνηση θα εγγυηθεί το 75% του περιεχομένου αυτού του χαρτοφυλακίου. Η κοινοβουλευτική έρευνα θα χρειαστεί περίπου 12 μήνες. Αυτά ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πράδος, ευχαριστούμε κύριε Ντερίκ. Άριστη παρουσίασή σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά που κάνετε στην Ολλανδία και στο Κοινοβούλιο. Πρόσφατα εγκρίνει την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια και έχετε και το διάλογο, έχουμε και το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ερωτήσεις και απαντήσεις με τον κύριο Ντεβίτ. Τρεις ερωτήσεις κάθε φορά. Αρχίζουμε με την κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, παρουσίαση των εργασιών σας. Εσείς μόλις όμως έχετε διοριστεί, διότι στην Επιτροπή μας όπου είχα εισηγήτρια, ήμουν εισηγήτρια εγκρίναμε μια ενδιάμεση έκθεση στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία και ο στόχος μας είναι αυτό το οποίο εσείς προτείνατε σήμερα να δούμε δηλαδή ποια είναι η αξιολόγηση στα διάφορα κράτη-μέλη και να μπορέσουμε να δράσουμε διασταυρωμένα. Εγώ δεν θα σας παρουσιάσω σήμερα τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε να σας το παρουσιάσουμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η δική μας εντολή ήταν πολύ ευρύτερη από τη δικιά σας, διότι το αντικείμενο της έρευνάς μας ήταν να εξετάσουμε τη χρηματοπιστωτική, την οικονομική και κοινωνική διάσταση της κρίσης. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα πεδίο υποβολής προτάσεων σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που έχετε εσείς. Τώρα, εσείς λέτε ότι ο καθοριστικός παράγοντας στις ρίζες της κρίσης είναι η, αγορά, η αμερικανική αγορά κινήτων. Αν εμείς κάνουμε μία τέτοια ανάλυση όμως, Και για να μην επαναληφθούν και πάλι αυτά, διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε ένα σπέκτρο, ένα παιδί πλαίσιο επιλογής ιδιαίτερα ευρύ. Η αγορά κινήτων, τον είπα, βασίζεται σε ένα μοντέλο που χρηματοδοτείται από το, από τα δάνεια, από ένα σύστημα που ζει με τα δάνεια. Και έστω και αν δεν το αποδείξαμε, δεν καταφέραμε να το αποδείξουμε, να το τεκμηριώσουμε ουσιαστικά, εγώ είμαι πάντα πεπισμένη ότι στην Αμερική το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί θέλησαν να πουλήσουν με δάνεια σπίτια σε ανθρώπους οι οποίοι κέρδισαν λιγότερα λεπτά. Αντίθετα με την Ευρώπη. Τώρα, μερικές ερωτήσεις για την Ολλανδική εμπειρία που πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται παραδειγματικά. Μιλήσατε εσείς ε, για τις προκλήσεις της ε, εύνομης διακυβέρνησης ότι δεν Είπαμε ακόμα το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα χρηματοπιστωτικά, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνο για τον, για για τον περιορισμό, για τη μείωση των πόνους, για τους υπαλλήλους, για τους μισθούς, για τη βαρύτητα των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, η δυνατότητα ψήφου με δανεικές μετοχές κλπ. Λοιπόν, τι διαπιστώσατε εσείς όμως και μετά για τις ε, καλές ε, και τις πρακτικές και τις λάθος πρακτικές για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Θεωρούνται οι κατοχώρες ως ε, παράδειγμα εύνομης διαχείρισης είναι υποχρεωτική η, συμμετοχή, η εγγραφή σε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο και ένα άλλο μοντέλο στην Ολλανδία είναι το μοντέλο εποπτείας. Πολλές φορές λοιπόν αναφέρθηκε το Ολλανδικό μοντέλο Twin Peaks ως παραδειγματικό. Τώρα η κρίση αμφισβητεί αυτό το μοντέλο. Αν το αμφισβητεί πραγματικά για μας δεν είναι ένα σοκ. Τώρα για τους ε, οργανισμούς ε, βαθμολόγησης ε, των του χρέους. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας εθνικός οργανισμός που να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είπατε όμως τίποτα για την φύση των κανόνων που διέπουν τους οργανισμούς Δέλτα Λάμδα Μιλήσατε επίσης και την οδηγία 2007 για το takeover στο τραπεζικό τομέα. Γιατί δεν έχει μεταφερθεί στο Ολλανδικό Δίκαιο. αφού ήδη το είχατε συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερές. Ο κύριος Θωμάς Μαν και μετά ο Όλε Σμιτ. Στη σειρά που ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντεβίτ, είπατε ότι ήσασταν ίσως υπερβολικά εξονυχιστικός. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε όλα αυτά τα τόσο σημαντικά μηνύματα από, από εσά. Είπατε ότι οι κοινοβουλευτικοί είχαν μονάχα περιορισμένε δυνατότητε να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα το θυμούνται όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό ισχύει και για τι ε, κάτω χώρε αλλά και για άλλου χώρου. Αλλά υπάρχει πάντα δυνατότητα παρέμβαση όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση. Όλοι θέλουν να δράσουν τότε. Και τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι και όχι να αφήσουμε σε κάποιους άλλους να αναλάβουν τα ίνια. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για εσά, για τις κάτω χώρες, και, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουμε μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και να επηρεάσουμε τις μελλοντικέ ε, ε, εξελίξεις χωρίς να καθυστερήσουμε και να έχουμε μια άλλη κρίση. Και είναι πολύ θετικό αυτό που είπε η δεύτερη βουλή των κάτω χωρών, ότι θέλουμε ένα σαφές σύστημα και διαφάνεια. Θέλω να σταθώ τώρα στο εποπτικό σύστημα. Είναι άτομα τα οποία πολλές φορές έχουν ε, πολύ καλές αμοιβέ, αλλά δεν ασκούν πάντα τον έλεγχο που πρέπει να είναι. Και είπατε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν καταστάσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν στρεβλές ακόμα και παραποιημένες πληροφορίες και στοιχεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Όχι μονάχα γιατί οι τράπεζες εξακολουθούν να επιμένουν σε ένα σύστημα αυτορυθμίσης, εγώ νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα σύστημα αξιόπιστο αν υπάρχει πραγματικός έλεγχος και όχι ένα σύστημα το οποίο οι τράπεζες για το δικό τους συμφέρον μπορούν να το διαστρέψουν και να το παραποιήσουν. Δεν είναι μονάχα λοιπόν το θέμα να αντιμετωπίσουμε βραχυπρόθεσμα την κρίση και μετά να γυρίσουμε στο business as usual. Όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουν τι απαραίτητε αρμοδιότητες και εξουσίες αυτά τα εποπτικά συμβούλια για να παρεμβαίνουν. Επίσης ένα άλλο ερώτημα. Είπατε, είχατε τη δυνατότητα να έχετε άμεσες μεταφορές πιστώσεων. Νομίζω ότι αναφερθήκατε, αλλά ότι κάνατε, κάνατε και άμεσες παρουσιάσεις μέσω της τηλεόρασης των συζητήσεων που έγιναν στην, ε, <clears throat> στην Επιτροπή σας και σε άλλες χώρες όπως το Βέλιο. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται με μικρές μονάχα εκπομπές, γίνεται με πιο εκτενείς ε, παρουσιάσεις στην τηλεόραση. Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί και εμείς θέλουμε στην Επιτροπή μας να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα θέματα αυτά. Και έρχομαι τώρα στο θέμα των, ε, της γερμανικής εμπειρίας. Υπάρχει αυτή η πρόταση στο Βερολίνο οι τράπεζες να δίδουν κάποιο ποσό το οποίο θα τροφοδοτήσει ένα ταμείο εγγύησης στο μέλλον. Τι πιθανότητα βλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο στις κάτω χώρες για να υπάρξει ένα τέτοιο μέτρο. Εμείς θεωρούμε ότι εάν προχωρήσουμε εμείς σε ένα τέτοιο σύστημα, ενώ οι υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης δεν συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι ένα μειονέκτημα για μα. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει αυτό και σε άλλες χώρες, λοιπόν. Και επίσης το σύστημά σας του Διοικητικού Επιτρόπου. Γνωρίζω ότι έχετε ένα σύστημα βάσει του οποίου υπάρχει ένας ombudsman, ένας διοικητικός επίτροπος, ο οποίος μπορεί να παρέμβει υπέρ των πολιτών και σε θέματα ε, χρηματοοικονομικά ακόμα. Υπάρχει ένα κεντρικό φορέα, ο οποίο παίζει αυτό το ρόλο του διαμεσολαβητή του διοικητικού επιτρόπου. Είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο και πώ μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό οι πολίτε. Τελευταίο και πιο δύσκολο ερώτημα. Είπατε ότι χρειάζεται ρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα εμείς ως Ευρωπαίοι να ε, να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε το πιστοτικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ελπίζουν ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικό, ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Ποια είναι τώρα η πιθανότητα να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό σε αρμονία και σε συνεργασία με όλο τον κόσμο, ότι ο Ομπάμα πράγματι θα κάνει τι απαραίτητε ε, μεταρρυθμίσει και στο δικό του σύστημα και ώστε μπορούμε επομένω να ρυθμίσουμε το πιστοτικό μα σύστημα χωρί να φεύγουν οι πιστοτικοί φορεί από την Ευρώπη και να πηγαίνουν κάπου αλλού που είναι πολύ πιο εύκολα. Και ξέρουμε ότι ορισμένα hedge funds έχουν φύγει αντισταθμιστικά κεφάλαια έχουν φύγει από, τα, από τις νήσους Καϊμάν αλλά αυτό δεν είναι παρά μόνο η απαρχή μια προσπάθεια να έχουμε περισσότερη διαφάνεια από ό,τι στο παρελθόν. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σμιτ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις κύριε Ντεβίτ. Ελπίζω να έχετε καλή μνήμη. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Εγώ είμαι Σουηδός και παραξενεύτηκα λιγάκι. Είμαστε από τους νόφερτους εμείς. Οι, οι ιδρυτές της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας απέτυχαν όταν εμφανίστηκε η κρίση. Γίνονται τόσο εθνικιστές ο καθένας από εσά στις χώρες Μπενελούξ. Πώς έγινε αυτό. Εμείς συνεργαζόμαστε στις βόρειες χώρες και προσπαθήσουμε να το λύσουμε το θέμα αυτό χωρίς την Ένωση. Με παραξένευσε αυτό. Θα ήθελα τα σχόλιά σας. Αυτή είναι η ουσία της Ένωσης, να μην είστε εθνικιστές, ακόμα και όταν πρόκειται για λεφτά. Δεύτερο, η iSafe Βρέχουμε από τον βορρά και η καρδιά μου χτυπάει για την Ιρλανδία. Και δεν ήταν μόνο η κατάρρευση της Αϊσεβ. E ήταν η κατάρρευση της Ισλανδίας που εξακολουθεί. Να δούμε εδώ τη σύνοψη. Καλό είναι ότι φέρετε κι εσείς μερική ευθύνη για την Ολλανδία. Γιατί αυτό στη συζήτηση δεν τονίστηκε, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα εγώ. Έχουμε και μερικού άλλου εδώ από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια χώρα 300.000, ε, όσο περίπου η πόλη από την οποία προέρχομαι. Και αν θέλει να επιζήσει αυτή η χώρα, πρέπει να του βοηθήσετε, κύριε Ντεβίτ. Και οι όροι που βάζετε στους πολίτες αυτούς που ακόμα ζουν σε αυτό το μικρό νησί και προσπαθούν να επιβιώσουν γιατί οι άλλοι θα φύγουν. Θα πάνε στην Αγγλία, στις σκανδιναβικές χώρες ή στην Ολλανδία για να βρουν εκεί το μέλλον τους και να δημιουργήσουν ενδεχομένω και άλλα προβλήματα για την Ισλανδία. Εγώ ελπίζω να φροντίσετε να ελαφρύνετε λίγο αυτούς τους όρους. Άκουσα φήμες που λένε ότι Ολλανδοί πολιτικοί θέτουν όρους στην συμμετοχή της Ισλανδίας στην Ένωση. Το θέμα της ISAF αν δεν λυθεί δεν θα γίνεται δεκτή στην Ένωση. Ελπίζω να το διαψεύσετε αυτό. Αυτές ήταν οι δύο ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για τα ενδιαφέροντα σχόλια και ερωτήσεις. Ο κύριος Δεβίτα έχει το λόγο να απαντήσει. Ehm, ehm, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με ερώτησαν. Ερωτήσεις ιδιαίτερα εύστοχες και σας ευχαριστώ για αυτές. Ευχαριστώ λοιπόν που με ρωτήσατε και αυτή ήταν η πιο απλή απάντηση που μπορούσα να δώσω. Τώρα, για την κυρία Μπερές. Εμείς ε, διαπιστώσαμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες βρίσκεται η βασική αιτία της κρίσης. Εξού δηλαδή και η παγκοσμιοποίηση της κρίσης, κρίσης ε, μέσα στην οποία ακόμη βρισκόμαστε. Εσείς το εξηγήσατε, γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση της αγοράς ακινήτων στις Ηνωμένε Πολιτείε, ποια είναι η κατάσταση στον δανειοδοτικό τομέα. Ο ανεύθυνος τρόπος χορήγησης δανείων σε ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να τα εξοφλήσουν, ε, αυτά είναι γεγονότα. Η πτώχευση της Lehman Brothers βρίσκεται επίσης στη ρίζα της κρίσης. Και εμείς Ολλανδοί δεν μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις στους ε, Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι πρέπει να τα ρυθμίσουν μόνοι τους αυτά που συμβαίνουν στη χώρα τους. Μιλήσατε επίσης για διαχείριση, για εύνομη διαχείριση κυρία Περές για τη συμμετοχή των εργαζομένων, για το μισθολογικό. Και αυτός είναι και ο μύτος της Αριάδνης που ενώνει πολλές από τις απορίες που εκφράζεται εδώ. Αυτό όμως δεν, αυτό όμως δεν εντάσσονται στη δική μας εντολή. Εμείς είχαμε ως εντολή να δούμε πως έχει η κρίση, όχι να μελετήσουμε τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Εμείς είδαμε ότι το δικό σας πεδίο διερεύνησης ήταν μεγαλύτερο από ότι το δικό μας. Η δική μας εντολή ήταν σαφώς πιο περιορισμένη. Μόνο τις επιπτώσεις της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί? Γιατί είμαστε μία μικρή επιτροπή στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Και εκπροσωπούνται 8 πολιτικά κόμματα σε αυτήν την επιτροπή. Μπορείτε να φανταστείτε κυρία μου ότι σε αυτήν την Επιτροπή υπάρχουν διεστάμενες απόψεις και γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή μας δεν είχε την αρμοδιότητα ούτε την εντολή να διερευνήσει ζητήματα τα οποία αφορούσαν σε άλλες επιτροπές. Τώρα για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Εμείς δεν θελήσαμε να επιστήσουμε, την, να, εξετάσουμε σε βάθος μάλλον αυτό το θέμα γιατί και την κοινή γνώμη δεν την ενδιαφέρει πολύ. Γιατί σε επίπεδο συνταξιοδοτικών ταμείων και εκεί υπάρχει η ίδια τάση ρίσκου στις επενδύσεις, αντίστοιχα με τις τράπεζες δηλαδή οπότε είχαν υποτιμήσεις. Εμείς ε, εξετάζουμε ιδιαίτερα σήμερα το θέμα της φερεγγιότητας των ε, ταμείων και η Ολλανδική Τράπεζα πρότεινε ορισμένα από αυτά τα ταμεία να αναλάβουν δρακόντια μέτρα και λόγω δηλαδή του κινδύνου που διατρέχουν θα πρέπει ίσως να σταματήσουν και να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες. Αυτό βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το συζητάμε. Το μέτρο, τα μέτρα αυτά απορρίφθηκαν μένα από το Κοινοβούλιο. Αυτό το μέτρο δηλαδή που ήθελε να επιβάλλει στα συνταξιδοτικά ταμεία ορισμένα μέτρα. Δεν θα ισχύσει λοιπόν αυτό το μέτρο. Διακόπτη κυρία Περές. Μήπως θα πρέπει να υποχρεωθούν τα τα ταμεία να έχουν μια μακροχρόνια στρατηγική επενδύσεων και να έχουν μια συγκεκριμένη δομή των χαρτοφυλακίων τους. Το πρόβλημα με κάτι τέτοιο, με μια τέτοια ρύθμιση, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι ότι δεν είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στα συντοξιδοτικά ταμεία και χωρισμένα. Κοιτάξαμε ποια είναι η σχέση των ταμείων αυτών με την πιστοτική κρίση. Στο βαθμό που υπάρχουν συνδέσεις, φυσικά το σχολιάσαμε στην έκθεσή μας, αλλά αυτό που αναφέρεται είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα από τους όρους αναφοράς της Επιτροπής μας. Λυπάμαι λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω περισσότερες περισσότερα στοιχεία και μορφή απαντήσεως. Αναφερθήκατε στο λεγόμενο μοντέλο Twin Peaks. Δίδυμε κορυφέ. Εμείς χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η ιδέα να έχουμε δηλαδή μια χωριστή λειτουργία της κεντρικής τράπεζας από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό είναι το μοντέλο. Τώρα είπαμε βέβαια ότι μετά από αυτά που έχουν γίνει, ίσως θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμε αυτό το το υπόδειγμα των Twin Peaks, δηλαδή χωριστή λειτουργία, για να δούμε αν είναι όλοι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει στην πράξη. Και αυτή είναι μια ιδέα που το Ολλανδικό Κοινοβούλιο υποστηρίζει. Γνωρίζετε ότι έχουμε τώρα μια νέα κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει την εξουσία πρόσφατα και ελπίζουμε όλοι ότι θα το θέσει και στην ημερησία διαταξή της νέα αυτή κυβέρνηση στις κάτω χώρες οργανισμοί πιστοληπτικής ε, βαθμολόγησης. Τι μπορώ να πω για αυτούς τους οργανισμούς. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι αυτοί οι φορείς βαθμολόγησης εκφεύγουν τις εποπτείες και πολλές φορές παίζουν διπλό ρόλο. <clears throat> Από τη μία πλευρά είναι φορείς που παρέχουν συμβουλές στις επιχειρήσεις και στις, στα χρηματοτραπεζικά ιδρύματα, ενώ συγχρόνως πολλές φορές <clears throat> συνεργάζονται ή λειτουργούν προς, σε, ως ε, εντολοδόχοι αυτών των ίδιων επιχειρήσεων και τραπεζικών ιδρυμάτων σε άλλα επίπεδα. Επομένως, Εδώ δεν έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, απλώς είπαμε ότι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να υπάγονται και αυτοί και αυτοί οι φορείς σε έλεγχο από τις εποπτικές αρχές. Γνωρίζουμε τις προτάσεις που αναφέρατε, αλλά δεν έχουμε εκφέρει άποψη λεπτομεριακά για τα θέματα αυτά. Τα λογιστικά πρότυπα επίσης. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι οι κανόνες λογιστικής λειτουργήσαν με υπερκυκλικό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις. Και επομένως, παράλληλα με την αύξηση των κεφαλουχικών απαιτήσεων στις τράπεζες, νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις ώστε να κάνει κανείς ένα κομπόδεμα για τις εποχές των ισχνών αγιλάδων. Δηλαδή θα πρέπει να λειτουργούν οι κανόνε αυτοί με έναν τρόπο αντικυκλικό και όχι υπερκυκλικό. Να μπορεί κανεί να δημιουργεί αποθέματα όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά στην άνοδο του οικονομικού κύκλου για να είναι έτοιμο κανεί να αντιμετωπίσει τι δύσκολε στιγμέ που έρχονται στη συνέχεια. Και πάλι για το θέμα της εποπτείας, εμείς πράγματι θέλουμε να έχει πιο διάφανο χαρακτήρα η εποπτεία για την οδηγία τον Βένετα. Ρωτήσατε γιατί εμείς δεν έχουμε μεταφέρει στο εθνικό μας σύστημα την νομοθεσία αυτή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο εξετάζεται από το Κοινοβούλιο των Κατοχωρών. Όπως σας είπα, λοιπόν υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά επειδή έχασε την εξουσία η προηγούμενη κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2010, και θεωρήθηκε αυτό ότι ήταν αμφιλεγόμενο νομοθέτημα, δεν το ε, υιοθέτησε η κυβέρνηση αυτή και πρέπει να επανέλθει η νέα κυβέρνηση. Ο στόχος της οδηγίας Αντών Βένετα ήταν ακριβώς να εξασφαλίσει ότι δεν υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και πολιτικοί παράγοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θεωρούμε όμως ότι ο έλεγχος της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Ολλανδικές αρχές όταν αξιολογούν την εξασφάλιση των απαραίτητων διασφαλίσεων σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Δεν διαβάζω πολύ καλά το όνομα σας. Α, Μαν λέγεστε. Ναι, κύριε Τόμας Μαν. Αναφερθήκατε στο θέμα των εποπτικών αρχών. Λέτε ότι δεν είχαν κάνει πολλά πράγματα οι εποπτικές αρχές και φυσικά ήταν αντικείμενο επικρίσεων για τον λόγο αυτό. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε εμείς βέβαια είναι ότι οι εποπτικές αρχές δεν κάνανε αρκετά πράγματα και όπως το λέμε στην εκθεσή μας, τίθεται εδώ πω ότι η κρίση θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια τροποποίηση του ρόλου των εποπτών, των εποπτικών αρχών. Πριν από αυτό, όπως μας είπαν οι πολλοί τραπεζίτες, ερχόντουσαν οι επόπτες στις τράπεζες, τους αντιμετωπίζαν με μεγάλο σεβασμό κτλ. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Έχουν πια περισσότερα εργαλεία οι εποπτικές αρχές, αλλά δεν είναι όλα προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα στο παρελθόν, αν ένας επόπτης έκανε κάποιες αυστηρές παρατηρήσεις σε μια τράπεζα, θα λαμβανόντουσαν υπόψη. Αλλά αυτό δεν γίνεται πια. Επομένω, χρειάζονται οι υπόπτε να έχουν περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή του και πρέπει να είναι και αυτοί πιο διάφανοι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δράσουν όταν αυτόν απαραίτητο χωρί να διστάζουν. Και θα πρέπει να αναλαμβάνουν δράση και όχι να φοβούνται επειδή μπορεί κάποιος να τους κάνει μια αστική αγωγή παραδείγματος χάρη λόγω των δρασεών τους. Οι εποπτικές αρχές λοιπόν και το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας μου επεξεργάζονται το θέμα αυτό και το Υπουργείο Οικονομικών έχει παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων <clears throat> που θα πρέπει να ε, δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα δράσης στις εποπτικές αρχές. και πιστεύω ότι πρέπει να λάβει χώρα και μια αλλαγή νοοτροπίας. Θα πρέπει να μπορέσουν να προσαρμοστούν <clears throat> στις νέες ε, συνθήκες και οι τράπεζες. Και τώρα έχουμε σε αυτό που είπατε για τις δημόσιες ακροάσεις, τις ε, εκπομπές που γίνονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που έγιναν αυτές οι συζητήσεις στο Ραδικό Κοινοβούλιο υπήρξε άμεση μετάδοσή τους από την τηλεόραση. Επίσης και στο ραδιόφωνο μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τις συζητήσεις. Και επίσης υπήρξε και σχολιασμός σε διάφορες ειδήσει για τα θέματα αυτά. Αλλά η τηλεόραση ήταν πάντα παρούσα στις συζητήσεις μας στο Κοινοβούλιο, στις ακροάσεις που κάναμε ως Επιτροπή για τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Το θέμα τώρα αυτό για τον λεγόμενο, για την ε, οικονομική συνεισφορά για από την πλευρά των τραπεζών. Και αυτό ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε, αλλά είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Όταν εμείς καταλήξαμε στην τελική μορφή της έκθεσής μας, διαπιστώσαμε ότι τελικά είχε εκφράσει θετική γνώμη για, ένα τέτοιο, για μια τέτοια εισφορά ή για ένα φόρο των τραπεζών το Ολλανδικό ε, Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά υπήρχε και μια ακόμα ιδέα για το τι μορφή θα έχει αυτή η εισφορά. Αν είναι ένα φόρο που ήδη υπάρχει, ή αν είναι κάποια ειδική εισφορά που θα θεσπιστεί. Και εδώ δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία στι κατοχώρε. Απλώ θα πρέπει, αν εφαρμοστεί μια τέτοια εισφορά, θα πρέπει να προσέξουμε και το να υπάρξει ισότητα ανταγωνισμού, δηλαδή να μην στρεβλώσει την, τον ανταγωνισμό η επιβολή αυτής της εισφοράς. Γι' αυτό του φόρου προς τις τράπεζες, και θα πρέπει να δούμε και ποια είναι και τα αποτελέσματα της συσσόρευσης όλων αυτών των μέτρων. Δηλαδή, ποια θα είναι η συνέπεια της συσσόρευσης όλων αυτών των μέτρων, τα οποία θα ρυθμίζουν εφ' εξής τον ε, τραπεζικό τομέα. Εμείς απλώς έχουμε περιορίσει την προσοχή μας στις προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν μια τέτοια εισφορά ή μια τέτοια φορολόγηση των τραπεζών. Για τον Ombudsman, όπως είπατε. επισήμως λέγεται διοικητικός επίτροπος ή διαμεσολαβητής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιος ε, εθνικός ε, επίτροπος διοικητικός, ο οποίος έχει ένα επιτελείο. Βέβαια είναι περιορισμένο το, το προσωπικό το οποίο στη διάθεσή του. Αλλά στην υπόθεση της Δέξια αυτός ο διοικητικός επίτροπος κατάφερε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. και φυσικά διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο για την εκπόνηση κανόνων και στην αντιμετώπιση διαμαχών σε σχέση με χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Είναι βέβαια εθνική φυσιογνωμία ο διαμεσολαβητής, αλλά είναι ένα άτομο, ένα πρόσωπο που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα Ε, διότι υπόκειται και στο, στην υποχρέωση απορρίτου, όπως όλες οι <clears throat> εποπτικές αρχές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θέλουμε λοιπόν <clears throat> να ισχύουν οι ίδιες ακριβώς ε, προδιαγραφές απορρίπτου όπως και για άλλες φορές. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι δεν έχει πάντα δυνατότητα να έχει στην, ε, στην κατοχή του όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητε για το έργο του. Και τώρα, <clears throat> για την, επί... Ε, για την δυνατότητα να έχουμε μια ρύθμιση η οποία θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Είναι γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο είχαμε μια χρηματοπιστωτική κρίση η οποία είχε παγκόσμιες επιπτώσεις. Θα έπρεπε λοιπόν και σε παγκόσμιο επίπεδο να εξευρεθούν οι λύσεις που θα αποτρέψουν μια τέτοια κρίση στο μέλλον. Η συνεδρίαση των G20, τα κράτη-μέλη των ε, G20, η Επιτροπή της Βασιλείας επίσης, έχουν αρχίσει να εργάζονται εδώ και αρκετό καιρό για να μπορέσουν να ρυθμίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Όλα αυτά βέβαια πηγαίνουν πολύ αργά. Συμφωνώ μαζί σας. Και σαν αποτέλεσμα θεωρούμε ότι αν κάποια στιγμή δούμε τα πράγματα πηγαίνουν πολύ αργά, ίσως θα πρέπει μόνοι μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουμε, αν δεν προχωρήσει σε επίπεδο παγκόσμιο. επί... σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακόμα και σε εθνικό επίπεδο να παίξουμε ένα ρόλο προδρόμων των G20, ιδίω σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει. Είναι μια ιδέα που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι ούτως ή άλλως τα επίπεδα των κεφαλοχικών ε, απαιτήσεων είναι πολύ χαμηλά και ο λόγος φερεγγιότητος θα είναι πολύ χαμηλός στις τραπεζές μας. Και στη συνέχεια το πακέτο Βασιλεία 3 προσπαθεί ακριβώς να αυξήσει το ποσοστό απεθεμάτων στο 9% με τα πρόσθετα μαξιλαράκια που θέλουμε εμείς να εισαγάγουμε. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι σίγουρα οι κάτω χώρες θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο περιθώριο λιγμών για να πάρουν τα μέτρα τα οποία θεωρούν επιδευλημένα. Αυτά λοιπόν για τα δικά σα ερωτήματα κύριε Μάν. Κύριε Σμίτ. Για τον Σουηδό φίλο κύριε Σμίτ. Αυτό που είπατε με, με ενδιαφέρει πάρα πολύ κύριε Σμίτ. Αυτό που είπατε για την Ευρώπη. Στη δεκαετία του 80 και εσείς Ζήσατε μια κρίση τον προηγούμενο αιώνα και μόλις, μόνοι σας βγήκατε από την κρίση με μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθεί πάντα μια εθνική λύση. Στη δεκαετία του 90 η κρίση που ζήσατε στην Σουηδία ήταν άλλου μεγέθους και άλλη μορφής από τη σημερινή. Δεν οφειλόταν στην παγκοσμιοποίηση, δεν ήταν μια παγκόσμια κρίση. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση. Τα τοξικά προϊόντα, τα τυκλοποιημένα προϊόντα όπως τα λέμε, κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Ε, το εμπόριο αυτών των προϊόντων. Αυτό δεν συνέβαινε στη δεκαετία του 90 η τιτλοποίηση πακέτων τίτλων μόλις ξεκινούσε τότε δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τότε κρίση σήμερα στην Ολλανδία έχουμε ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε εν μέρη εθνικά αλλά όταν βλέπουμε τη σχέση που υπάρχει με τον υπόλοιπο κόσμο διαπιστώνουμε ότι όλα είναι αλληλένδετα με την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου αργά ή γρήγορα πρέπει όσο γίνεται να βρίσκουμε παγκόσμιες λύσεις. Έστω και αν αυτό παραμένει εν μέρει ευχολόγιο. Και αυτό είπα και στον κύριο Τόμας Μαν. Αναφερθήκατε στην iSafe. Δύσκολο πρόβλημα αυτό για μας κύριε Σμιτ. Η Ολλανδία ως κράτος παρενεύει για να προστατεύσει τον καταθέτη το ποσό στο σύστημα εγγύσεων των καταθέσεων αυξήθηκε σε 100.000 ευρώ κατά καταθέτη. Το σύστημα εγγύσεων των καταθέσεων και η συνολική αναγκαία 1,3 δις που το έχουμε ως πίστοση Ολλανδία-Ισλανδία αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο της έρευνας στο δεύτερο σκέλος των εργασιών της Επιτροπής μας. Αν πω κάτι, θα ήταν σαν να προδίκασα τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης της έρευνάς μας, που μόλις τώρα ξεκίνησε. Το θέμα είναι ακανθόδες, λεπτό, στη σχέση μας με την Ισλανδία. Κάνετε και ένα άλλο ερώτημα. Είπατε είναι λογικό οι Ολλανδικές αρχές να δίνουν εγγυήσει στους πολίτες τους, να δίνουν λεφτά και μετά να προσπαθούν να πάρουν πίσω τα χρήματα αυτά από την Ισλανδία. Δεν θέλω να υπεκφύγω την ερώτηση, αλλά δεν ξέρω και αν μπορώ να απαντήσω. Θεωρώ ότι φρόνιμο ήταν να βοηθήσουμε τους καταθέτες μας και φυσιολογικό είναι να προσπαθούμε να ανακτήσουμε ένα τιμήμα αυτό που πληρώσαμε. Τώρα, η ερώτησή σας πιο γενική για την ένταξη της Ισλανδίας στην Ένωση. Είναι πολιτικό το θέμα αυτό. εξοχή πολιτικό. Και δεν έχει καμία σχέση με την εντολή για την έρευνα που κάνουμε. Δεν το συζητάμε αυτό εμείς καθόλου. Το σύστημα στην Ολλανδία προβλέπει μια επιτροπή στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Οικονομικών που συζητάει με τον Υπουργό για λόγους ασφάλειας για μη που πω πράγματα και μετανιώσω μετά λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας μετά από έναν χρόνο θα έχει εγκριθεί η εκθεσή μας ίσως τότε να είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτησή σας ελπίζω να μην ξέχασα καμία ερώτηση Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεβίτ. Απαντήσατε διαμακρών. Επόμενος γύρος. Αν οι, οι ερωτήσεις... Δεν ξέρω αν θα έχουμε ίσως λιγότερου ομιλητές. Αρχίζουμε πάση με την κυρία Βόρτμαν Κόλ. Αγγλικά. Ολλανδικά μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ συνάδελφοι. Σας αποκαλώ συνάδελφο, διότι πραγίστηκε εσείς από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι για το ότι ήρθατε εδώ σήμερα μια μέρα που θα πρέπει να μιλήσετε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, διότι εκεί γίνεται η συζήτηση για την, η συζήτηση για τη νέα κυβέρνηση. Ήταν ευγενές εκ που βρήκατε το χρόνο να έρθετε να συνδιαλεγείτε με, με Πρώτο, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Ρέφενεστα, η όρια αναφορά τη Επιτροπή σα στην Ολλανδία. Πολλά χρήματα των φορολογούμενων κατέληξαν σε τράπεζες. Στη χρηματοπιστωτική κρίση η Επιτροπή σας είχε την εντολή να διεξάγει αυτή την έρευνα Κατανοώ ότι είστε σε δύσκολη θέση να απαντήσετε στις δύσκολες ερωτήσεις του συναδέλφου Σμιτ Φερπίν. Εδώ είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο και οι ερωτήσει που σας υποβάλλουμε σαν να εκπροσωπείτε όλο το Ολλανδικό Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Κυβέρνηση ενώ εσείς είστε μέλος ενός κόμματος που είναι εδώ και καιρό στην αντιπολίτευση. Αυτό προκειμένου να οριθιτούνται οι θέσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Με παραξενεύει το γεγονός και παρακολουθώ τις εργασίες της Επιτροπής σας ότι οι έρευνές σας αφορούν κυρίως την κατάσταση στην Ολλανδία και οι συστάσεις σας κυρίως αφορούν κανονισμούς και λοιπά που αφορούν την Ολλανδική που θα πρέπει να τους ε, χειριστεί η Ολλανδική κυβέρνηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους εδώ εμπλεκόμενους φορείς περισσότεροι θα έλεγα ξεπερνάνε τα σύνορα. Σύνορα της Ευρώπης είναι παγκόσμιο χαρακτήρα. Το είπατε κι εσείς. Χρειαζόμαστε έναν κανονισμό. Με παραξενεύει λοιπόν το ότι το σχόλιο σας ότι χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο χαρακτήρα οργανισμό και αν όχι τουλάχιστον ένα εθνικό κανονισμό. Μήπως υποτιμάτε τη σημασία των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δεύτερο τμήμα των ερευνών σας εστιαστήκατε στην Ολλανδική κατάσταση μέχρι σήμερα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να, έχετε, να προσθέσετε μια ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτό. Δύο παραδείγματα για να δείτε ότι έχετε συμμάχους στο Ευρωκοινοβούλιο. Ανακαλύψατε ότι τα κράτη-μέλη σύντομα ξέχασαν την κρίση όσον αφορά συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάμε για την υποπτία των τραπεζών λέτε ότι χρειάζεται σκληρή εποπτεία. Αλλά το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών αποδυνάμωσε τις προτάσεις αυτές. Εμείς δεν θέλαμε να αποδυναμωθούν αυτές οι προτάσεις και γι' αυτό χάρη στο Κοινοβούλιο όμως, είχαμε πιο σκληρή νομοθεσία. Το ίδιο και για τα πριμ. Μιλάτε για τον τραπεζικό κώδικα, αλλά ξέρετε ότι όλοι οι φορείς στηρίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα τους αφορά ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο μηχανισμός επίλυσης της κρίσης, ένα δεύτερο παράδειγμα, και η τραπεζική εισφορά που συζητιέται. Και εδώ προσπαθούν να τον αποδυναμώσουν οι κυβερνήσεις. Εμείς θέλαμε μια γνήσια ευρωπαϊκή, ε, ευρωπαϊκό σύστημα. Για το σύστημα των καταθέσεων, εγγύησης καταθέσεων, η κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα. Εμείς θέλουμε ένα ευρωπαϊκό θα βοηθούσε να λυθούν τα προβλήματα. Το ίδιο ισχύει για καλύτερη μακροοικονομική εποπτεία. Έχει υποβληθεί ένα σχετικό νομοθετικό πακέτο και γι' αυτό. Και ρωτώ, έχετε επαφές με άλλες αντίστοιχες επιτροπές σε άλλα εθνικά κοινοβούλια να δείτε τι κοινά συμφέροντα υπάρχουν, να υπάρχει μια σκληρή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Και μια δεύτερη ερώτηση. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω από το να υποβάλλετε κανονισμού στην Ολλανδική κυβέρνηση. Σε σχέση να αναζητήσετε ευρωπαϊκές λύσεις. Στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο φαίνεται να μην υπάρχει αυτή η φιλοδοξία αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να αυξηθεί το επίπεδο συνειδητοποίηση, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτό το επίπεδο, πρόεδρος, ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεβίτ για όσα μας είπε, πολύ ενδιαφέροντα. Θα είμαι σύντομο στις ερωτήσεις μου. Αναφερθήκατε στο CRS, στις αξιολογικούς οίκους. Όταν η κυρία Μπέρες ήταν πρόεδρος στην Ελληνική Επιτροπή, οι οίκοι αυτοί, λόγω των δραστηριοτήτων, κάτι τους καλέσαμε να πούν. Δεν βλέπετε ότι οι ίδιοι οίκοι αξιολογούν κυβερνήσεις και οι αγορές ομολόγων αξιολογούν κυβερνήσεις. Δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας ρυθμίζει το δημόσιο τομέα. Αυτό το έχετε σκεφτεί. Υπάρχουν και κτημένα συμφέροντα εδώ στο παρελθόν ήταν δυνατόν να επιτραπεί αυτοί να αξιολογούν τι κάνει ο δημόσιο τομέα κυβερνήσει με βάση τι δικέ του επιδόσει στο παρελθόν. Δεύτερον, τα χαμηλά επιτόκια και ο έλεγχο του πληθωρισμού όσον αφορά τον πληθωρισμό στοιχείων ενεργητικών. Επί δύο χρόνια ερωτώ τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας στην Οικονομική Επιτροπή μας σχετικά με το θέμα της του πληθωρισμού των στοιχείων ενεργητικού. Στη χώρα μου, αν δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα του asset inflation, πληθωρισμού στοιχείων ενεργητικού, θα τα πηγαίναμε πολύ καλά. Επειδή έχουμε σε αυτό το πρόβλημα στην Ιρλανδία, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Τρίτη ερώτηση. Φτάσαμε εδώ που είμαστε, διότι σε μεγάλο βαθμό το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν λειτουργούσε με αυτοματισμούς, με συστήματα υπολογιστών κλπ. Ακόμα και στις τράπεζες ένας υπολογιστής αποφασίζει να στείλει μια επιστολή σε ένα πελάτη σήμερα. Σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, διάφορα όργανα αγόρασαν προϊόντα που δεν καταλάβαιναν. Είχαν τρία αλφα τα προϊόντα αυτά και μέσα είχαν τα περίφημα subprime, τα τοξικά. Έχω άλλη μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν αφορά την Ολλανδία. Σίγουρα αφορά την Ιρλανδία. Και δεν μιλάω για την μεγάλη εικόνα. Αν βγούμε από την κρίση, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια θέση απασχόλησης κατά μικρή, μικρομεσαία απασχόληση που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας σε όλες τις χώρες, όταν είχαμε στο παρελθόν διευθυντέ γραφείων τραπεζών, γνωρίζανε τον πελάτη του, γνωρίζανε πώ θα πάει, πώ λειτουργεί, τι επιχειρησιακό μοντέλο έχει. Αυτό ισχύει για τη χώρα μου. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στους κλασικούς διευθυντές τραπεζών που πάβουν να παίζουν σαν να παίζουν σε καζίνο και να υπολογίζουν και να λαμβάνουν σταθμισμένους κινδύνους. Γιατί αν δουλεύουν μόνο για το κέρδος, ένας ένας κόσμος θα τρέχανε στην αγορά. Όχι καζίνο όχι να παίζουν παιχνίδια, όχι αυτομετωπιμένα προγράμματα μέσω υπολογισμών άτομα που να κρίνουν με βάση το χαρακτήρα, τις επαγγελματικές επιδόσεις, κλασικούς τραπεζ, ε, διευθυντές τραπεζών. Το έχετε σκεφτείτε αυτό. Ευχαριστώ και πάλι για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ένα ερώτημα από την κυρία Φόρτ. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος ε, ομιλητής. Σίγουρα, αν ο δημόσιος τομέας δεν ζητούσε από τον ιδιωτικό τομέα να δανείζει χρήματα, δεν θα χρειαζόταν και επιχείρηση διάσωση στη συνέχεια. Εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια που κάνατε για την κατάσταση των κάτω χωρών και νιώθω μεγάλη κατανόηση και συμπαράσταση για αυτά τα οποία αναφέρατε. Είπατε ότι σε εθνικό επίπεδο υπήρχαν λήπτες αποφάσεων που είχαν τις εξουσίες και θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν για να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά για κάποιους λόγους αποφασίσαν να μην χρησιμοποιήσουν αυτές τις εξουσίες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είδαμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτι το οποίο θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Δύο ερωτήσεις. Είπατε για πιο υπεύθυνου μετόχους. Κάτι το οποίο έχουμε τονίσει και εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ζητήσατε επίσης να υπάρχει και πιο υπεύθυνη λογιστική μέθοδος. Μπορείτε να μας πείτε για το ρόλο των μετόχων και πώς μπορούν να δρουν με πιο υπεύθυνο τρόπο και για το θέμα της λογιστικής είπατε ότι η λογιστική απογραφή θα πρέπει να δίνει σαφή εικόνα των κινδύνων στους ετήσιους λογαριασμούς. Έχετε σκεφτεί αν οι λογιστές θα πρέπει να είναι παρόντες στα συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, αν θα πρέπει να είναι παρόντες στα διοικητικά συμβούλια, μήπως θα, έχουν, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια αστική ευθύνη ε, ως ε, οικονομικοί ελεκτές όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Δεν είναι Βλέπω, λέει ο κύριος ε, Μίτσελ, ότι ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα αυτορυθμίζεται. Εμείς θα πρέπει να ρυθμίσουμε, αλλιώ δίνουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν προβεί σε καταχρήσεις στο παρελθόν να το δικαίωμα να ρυθμίσουν τα δικά τους όπω θέλουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ήταν στο παρελθόν με τους δημόσιου φορείς. Υπήρξαν και συγκρούσεις συμφερόντων ακόμα, αλλά θέλω να υπάρχει κάποιο φορέα στον οποίο να μπορούμε να εμπιστευόμαστε επιτέλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Ντεβίτ. Χωρίς μικρόφωνο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία κολ ε, έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Με ρωτήσατε, μα τι στο καλό κάνεις εδώ ενώ έπρεπε να είσαι στην Ολλανδία. Καταλαβαίνω λοιπόν πολύ καλά ότι εκτιμά την παρουσία μου στο χώρο. Πράγματι, δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό, θα αντισταθώ μάλλον στον πειρασμό να κάνω τουρισμό στις Βρυξέλλες διότι πρέπει να τρέξω γρήγορα πίσω. Καλά κάνατε που μου το θυμήσατε για το πού πρέπει να βρίσκομαι. Για να συνοψίσω την τοποθέτησή σας εσείς ε, μου καταλογίζετε μας καταλογίζεται ότι δεν λάβαμε υπόψη μας επαρκώς την ευρωπαϊκή πτυχή. Εμείς φυσικά και λάβαμε υπόψη μας και την ευρωπαϊκή πτυχή και το διεθνές επίπεδο, την Βασιλεία, το G20 και στη βάση λοιπόν των εμπειριών μας μπορούμε να πούμε ότι απαιτούμε, θεωρούμε απαραίτητη μία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα θέλαμε να ξεπεράσουμε και αυτό το τριπλό σύστημα το οποίο προτείνει η ομάδα Λαροζιέρ. Θέλουμε να μας δοθεί δυνατότητα να λάβουμε και μέτρα αν χρειάζεται. Μετά. Δεν ξέρω αν εσείς ή κάποιος άλλος μου το ρώτησε, αλλά υπόθηκε ότι τα συστήματα διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Τώρα, στη βάση της συμφωνίας iSafe, διαπιστώσαμε ότι θα έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα με φορολόγηση που να συνδέεται με την επικινδυνότητα των επενδύσεων. Τώρα για τη φορολόγηση των τραπεζών είπαμε πρέπει να παρέμβει η Ευρώπη και ο υπουργό μας ήδη έχει εκφραστεί και πολύ πιθανώς να ισχύσει στις κάτω χώρες αυτού του είδους η φορολόγηση. Αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει ρύθμιση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως γνωρίζουμε ότι επίγει η επίλυση του προβλήματος. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και εκείνη η αίσθηση συγκράτησης και μετριοπάθειας. Δηλαδή θέλουμε η δράση να είναι μελετημένη για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά και να λειτουργήσει το σύστημα. Αν εμείς λοιπόν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να κινηθεί κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο, ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε και ο υπεύθυνο της, ε, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ολλανδίας είπε ότι θα δράσουμε μονάχοι μας διότι οι υπόλοιποι κολλησιεργούν. Η παρέμβαση ήταν κατεπίγουσα, δεν μπορούσαμε λοιπόν να περιμένουμε. Αν μπορώ να παρεύω μια στιγμή κυρία Πρόεδρε, να κάνω ένα σχόλιο. Στα Ολλανδικά το κάνω. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε πολύ καλά. Αυτό όμως το οποίο προσπάθησα να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναφέρεται στην έκθεση Τελαροζιέ ή για άλλα εγχειρήματα αυτού του είδους θέλει να υλοποιήσει αυτό το οποίο ζητάτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δικό μας κοινοβούλιο σας υποστηρίζει πλήρως, αλλά υπάρχει μια τάση από τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια να μην ακολουθούν αυτή την κίνηση. Εσείς έχετε επαφή με άλλα εθνικά κοινοβούλια. Μήπως θα πρέπει και τα άλλα εθνικά κοινοβούλια να σας βοηθήσουν για να πετύχετε αυτούς τους στόχους και αυτές τις φιλοδοξίες. Κάτι το οποίο ήταν πολύ καλό για τις χώρες. Είχαμε επαφές προφανώς με το Βελικό Κοινοβούλιο καταρχήν. Δύο επιτροπές ήτανε αρμόδιες για αυτό το ντοσιέ στο Βελγικό Κοινοβούλιο και ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Αλλά λόγω της κυβερνητικής κατάστασης στο Βέλγιο δεν ευόδωσε η συνεργασία. Ο πρόεδρος της ε, Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας επειδή ακριβώς ασχολιόμασταν με την κρίση θέλησε και θέλει και το επαναλαμβάνει ότι πρέπει να υπάρχει διεθνής διαβούλευση, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τα άλλα εθνικά κοινοβούλια τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Ως Ερευνητική Επιτροπή όμως εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα, εμείς επαφές μπορούμε μόνο να έχουμε Τώρα να σταθώ και στα άλλα θέματα. Ψάχνω τα ντοσιέ μου. Ανάτο. Λοιπόν, να σας μιλήσω για το καθεστώς εγγύησης καταθέσεων. Κυρία Μίτσελ, α όχι, κύριος Μίτσελ, καλά κάνατε και με διορθώσατε, περί κυρίου πρόκειται. Λοιπόν, εσείς μιλήσατε για τους ε, οργανισμούς ε, εκτίμησης. Και μιλήσατε επίσης και για το αυτοματοποιημένο σύστημα σε τραπεζικό επίπεδο. Εμείς εξετάσαμε πολύ καλά το ντοσιέ και όταν εξετάσαμε και το iSafe και το ντοσιέ της τράπεζας DSB διαπιστώσαμε ότι το internet banking η αυτοματοποίηση και η ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Κρήτη. Διότι όλα γίνονται στιγμιαία. Όχι όπως στο παρελθόν που κάποιος έκανε δύο μέρες ουρά έξω από την τράπεζα. Πρέπει λοιπόν εμείς να δημιουργήσουμε και πάλι κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζίτη και καταναλωτή. Να έχουμε έναν τραπεζίτη που να ξέρει τι προϊόντα πουλάει. Έχουμε την Αμπένα Άμρο στην Ολλανδία διαπιστώσαμε ότι με την παλιά δομή είχαμε τον αρμόδιο που παρουσίαζε το προϊόν ένα προς ένα και στον τραπεζίτη που μετά το πουλάγε στον καταναλωτή σήμερα πουλάνε πακέτα, package και δεν ξέρουν τι πουλάνε μέσα. Και ο αρμόδιος λοιπόν για αυτά τα πακέτα δεν ήξερε από τι το πακέτο, αποτελούταν το πακέτο. Ήταν κάτι το ακατανόητο. Αυτό σημαίνει τεράστιο ρίσκο. Χρειάζεται λοιπόν μία διαχείριση του κινδύνου, έλεγχος του κινδύνου και αξιολόγηση του κινδύνου. Πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο. Και αυτή η διαχείριση λοιπόν του κινδύνου πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του τραπεζικού κώδικα. Δεν έγινε ακόμα αλλά πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτός ο κώδικας. Είναι <coughs> μία πρόταση αυτορύθμισης των τραπεζών. Αλλά εμείς είπαμε ότι αν δεν υπάρξει μία καλύτερη αξιολόγηση δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να παρέμβουμε. Δηλαδή οι τράπεζες μονάχες τους δεν μπορούν να αυτορυθμιστούν. Κυρία Φόρντ, ένα λεπτό. Καταρχήν. Έχετε δίκιο κυρία Φόρντ. Πολύ σωστά το είπατε. Οι μέτοχοι τη θέση του. τους. θέλουν πάντα μεγαλύτερα κέρδη οι μέτοχοι. Όχι μόνο ενίσχυση του μετόχου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο θέλει και return, θέλει επιστροφή. Ο μέτοχος πλέον βλέπει βραχυπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα. Θέλει να έχει άμεσο μέρισμα, άμεσα κέρδη. Και αυτό εις βάρος επιχείρησης. Αυτό λοιπόν εμείς που προτείναμε για να καταπολεμήσουμε αυτήν την τάση είναι οι μέτοχοι να εμπλέκονται περισσότερο μέσα στη διαχείριση του, της τράπεζας. Πώς. Όταν ένας μέτοχος κρατάει περισσότερο καιρό τις μετοχές του χωρίς να τις ρευστοποιεί, τότε η ψήφος του θα βαραίνει περισσότερο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή πιο πολύ τα λεφτά σας είναι δεσμευμένα σε μετοχές, τόσο μεγαλύτερη θα και η επίδρασή σας στη δίκη στον επιχείρησης. Αυτό προτείνουμε τώρα για τις ετήσιες εκθέσεις. Τι εστί η αιτήσια έκθεση. Πρόκειται για ένα τούβλο, για έναν τόμο τεράστιο. Που φτιάχνουν, το γράφουν οι λογιστές. Και να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των λογιστών μέσα αυτή την κρίση. Όχι μόνο δηλαδή για τις τράπεζες, αλλά και για τις ασφάλειες. Για την τάση. Είπαμε ότι οι λογίστες θα πρέπει να αναλαμβάνουν και την εκτίμηση του κινδύνου και την παρακολούθηση της αγοράς. την ΑΕΘΕΜ αλλά και άλλες επαγγελματικές ρώσεις. Και ήρθαμε σε επαφή λοιπόν με όλες αυτές τις οργανώσεις των λογιστών <coughs> οι οποίες μας ρώτησαν τι θέλαμε και τους είπαμε εμείς λογιστικές εκθέσεις που να βελτιώνουν την ετήσια έκθεση μιας επιχείρησης διότι αυτή η έκθεση αποτελεί βάση πληροφόρησης για έναν τρίτο μελλοντικό επενδυτή. Πρέπει λοιπόν ο λογιστής να είναι αξιόπιστος όταν κάνει την έκθεση όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και έναντι των επενδυτών. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι σχεδόν παντού στον κόσμο, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, ο κύριος Γκρίνσπαν ήταν αυτός που άσκησε κυρίως αυτή την πολιτική. Στη μείωση των επιτοκίων. Δηλαδή την πολιτική του ιστορικά χαμηλότερου τόκου. Και αυτό δηλαδή <coughs> για να διασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη. Ο Άλαν Γκρίνσπαν έκανε λάθος. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν σωστή αυτή η πολιτική. Και έπαιξε ρόλο στην κρίση των subprimes αυτή η πολιτική. Και οδήγησε δηλαδή και στην κρίση που γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σα, κύριε Στογιάν. Τώρα έχετε και εσείς το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση μόνο. Στην ανάλυση αυτή που κάνατε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο λάβατε υπόψη και τη συμπεριφορά των Ολλανδικών τραπεζών στις αναδυόμενες οικονομίες. συμπεριλαμβανομένη και της χώρας μου της Ρουμανίας όπου η χρηματοπιστωτική κρίση δεν καθορίστηκε τόσο από τα τοξικά προϊόντα και επενδύσει, όσο από το ότι δόθηκε μια πληθώρα καταναλωτικών πιστώσεων όχι μόνο οι Ολλανδικές τράπεζες και οι Αυστριακές τράπεζες και άλλες έδωσαν αυτά τα χρήματα μια χιονοστιβάδα καταναλωτικών πιστώσεων. Και όταν ήρθε η κρίση, σταμάτησε η ρευστότητα και εμφανίστηκαν τα προβλήματα. Και ρωτώ, λάβατε υπόψη τη συμπεριφορά των Ολλανδικών τραπεζών στις χώρες αυτές και ποια ήταν η επίπτωση αυτής της συμπεριφοράς στα προβλήματα αυτά που ζήσατε μετά και στην Ολλανδία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεβίτ θα απαντήσει εφόσον κανένας άλλος δεν ζητάει το λόγο. Έχω κι εγώ μία ερώτηση για την εντολή της Επιτροπής σας. Όταν εμείς εδώ συστήθηκε η ειδική αυτή Επιτροπή, συνοψίσαμε τις αιτίε και τις συνέπειες της κρίσης, αλλά τελικά οι συστάσεις που θα δώσουμε δεν θα έχουν νομοθετική ισχύ, θα είναι μόνο συστάσεις προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Και ρωτώ, η δική σας εντολή ποια είναι είναι παρόμοιο τη δική μας ή θα έχει κάποια νομιμαθητική επίπτωση. Απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η στάση των ε, Ολλανδικών ομίλων μέσα στο πλαίσιο αυτό που διαγράψετε, εγώ γνωρίζω ότι πράγματι έχουν δώσει πολλές πιστώσεις οι Ολλανδικοί οι τραπεζικοί όμιλοι σε ορισμένες χώρες. Και γνωρίζω ότι σε κάποια χρονική στιγμή οι πιστώσεις αυτές ουσιαστικά σταμάτησαν απότομα, δηλαδή έκλεισε η βρύση. Αλλά αυτό έγινε και σε παγκόσμιο επίπεδο ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε το λεγόμενο credit crunch, δηλαδή σταμάτησε η παροχή πιστώσεων, υπήρξε μια απόλυτη έλλειψη ρευστότητος και αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα να οξύνει την κρίση. Και αυτό ίσχυσε και στην περίπτωση των κάτω χωρών ή κατοχωρήτικες τράπεζες χωρίς καμία αμφιβολία υπέστησαν και τις συνέπειες αυτές της πράξης. Αυτό δεν το εξετάσαμε για να μην ειλικρινείς. Δεν εξετάσαμε την συμπεριφορά των Ολλανδικών τραπεζών στις λεγόμενες από εσά αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες καλύτερα χώρες και δεν ήταν αυτό τμήμα και της εντολής μας. Αλλά για την ίδια την χώρα μας, για την Ολλανδία, στο Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών συζητήσαμε μαζί με την κυβέρνηση συζητήσαμε για τις συνέπειες της ε, διακοπής της παροχής πιστώσεων. Ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν οδυνηρά τα αποτελέσματα. Ήταν πολλές οι εταιρείε και οι ιδιώτες που αντιμετωπίσαν τεράστια προβλήματα και επομένως γνωρίζω το πρόβλημα που αναφέρεται. Απλώς εμείς σαν Επιτροπή Έρευνας δεν είχαμε εντολή να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συστάσεις σχετικά, αλλά δεν ήταν μέσα στην εντολή μας. Το μόνο το οποίο γνωρίζω ήταν ότι αυτό ήταν φυσικά ένα ευρύτερο πρόβλημα από το πρόβλημα των κατοχωρών. Και εμείς επλήγημεν από την έλλειψη πιστώσεων στην αγορά. Για το ερώτημα της κυρίας Προέδρου, <clears throat> σε σχέση με το χαρακτήρα των, των συστάσεων που θα μπορούσαμε εμείς να διατυπώσουμε. Θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει τις δικές μας συστάσεις με αυτές που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή σας. Μα υπάρχει μια πλειάδα συστάσεων που προέρχεται από τις δικές μας συστάσεις. Κάποιες από τις δικές μας συστάσεις έχουν ήδη μεταφραστεί σε πολιτικές αποφάσεις. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη, ενέκρινε ομόφωνα μια σειρά ρυθμίσεών μας και επομένως τις έχει μετατρέψει σε νόμους. Παραμένουν όμως άλλες συστάσεις μας που θα πρέπει να οδηγήσουν στην εκπόνηση νομοθετικών πράξεων. Κάποιε λοιπόν από αυτέ δεν έχουν περάσει επομένω στην Ολλανδική Ένωμη Τάξη. Παραδείγματο χάρη η νομοθεσία για την χρηματοοικονομική εποπτεία, ο κώδικς τραπεζών, όπου πρέπει να γίνουν ακόμα κάποιες ενέργειες, κάποιες ε, ε κάποια επεξήρεση. Ο θεματοφύλακας της αγοράς. Αν ξαναγυρίσουμε στην Αμπέν Αμρό. Τον Οκτώβριο του 2008 δεν υπήρχε κανένας Ολλανδικός νόμος ο οποίος να ρυθμίζει την ε, πρόταση εξαγοράς, τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΑΜΡΟ. Εάν υπήρχε θα μπορούσε να είχε παρέμβει ή να είχαν παρέμβει οι Ολλανδικές αρχές. Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία τα οποία εμείς προτείνουμε για τις εποπτικές αρχές των αγορών θα έπρεπε να έχουν σαν αποτέλεσμα μια τροποποίηση της Ολλανδικής νομοθεσίας. Και θα τροποποιηθεί η νομοθεσία αυτή. Έχουμε προτείνει πράγματι μια σειρά από εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα εγκριθούν από το Κοινοβουλίο μας, θα γίνουν νόμοι και όπως ξέρετε φυσικά η διαδικασία η νομοθετική είναι χρονοβόρα και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης είδαμε ότι οι λεγόμενες ανοιχτές πωλήσει, οι οποίες τώρα έχουν ε, απαγορευτεί, <clears throat> είχαν ε, παίξει μεγάλο ρόλο και είχαν χρησιμοποιηθεί σε ευρία κλίμακα. Το λεγόμενο short selling, οι ανοιχτέ πωλήσει, θα είναι εφ' εξής υποκείμενες σε μια ρύθμιση, σε κανόνες και τόνιζω, τονίζω και πάλι θέλουμε να συνεχίσουμε την δραστηριότητά μας και να ξεπεράσουμε το επίπεδο των συστάσεων. Θα ζητήσουμε τώρα από την κυβέρνησή μας, από το Κοινοβούλιο όμως μάλλον, να ελέγχει και την κυβέρνηση για να δει κατά πόσον αυτές οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο γίνονται πραγματικότητα και σε καθημερινό επίπεδο. Σαν Επιτροπή Έρευνα, ο στόχο μα είναι να διατηρήσουμε την αίσθηση του κατεπήγοντο για τη ρύθμιση για αυτά τα θέματα. Αυτό είναι ουσιώδε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την επανάληψη μια κρίση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Ντεουίτ. Κύριε Μπερέ, θέλετε να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων ήταν πολύ χρήσιμη για το δεύτερο τμήμα της εντολής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί γνωρίζω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν στη δική σας Επιτροπή ίσως όχι πάντα με την ίδια αποτελεσματικότητα έγιναν και σε άλλα κρατημέλη. <clears throat> και θα είναι χρήσιμο να δείτε τι ψηφίσαμε και εμείς με μεγάλη πλειοψηφία στην πρόσφατη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. αυτά που είπε η συνάδελφος η κυρία Βόρτμαν Κόλ η οποία είχε άλλες δεσμεύσεις για την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου το οποίο έχετε αναλάβει νομίζω και πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ κατέγραψα από αυτά που είπατε το ότι μιλήσατε και για το όριο, το κατόφλι των 100.000 ευρώ για την προστασία των καταθετών και την εγγύηση των καταθέσεων. <clears throat> Αυτό είναι τώρα ένα ευρωπαϊκό κατόφλι. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση και κοινή διάγνωση και νομίζω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία ώστε να δημιουργήσουμε μια συγκλίνουσα ε, δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο για αλληλοϊποστήριξη των ενεργειών μας και χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να γευματίσουμε μαζί και θα συζητήσουμε και για τα νομισματικά διακυβευόμενα τα οποία βέβαια εκφεύγουν λιγάκι από την εντολή που έχετε ως ε, Επιτροπή Έρευνας για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, αλλά που είχαν και πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλο ρόλο στη δράση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και με ενδιαφέρει πολύ αυτό που είπε η συνάδελφος για την πρακτική της Αμερικανικής του Αμερικανικού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και για το ρόλο που έπαιξαν σε ό,τι αφορά τις κερδοσκοπικέ δραστηριότητε. Σας ευχαριστώ πάντω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και βλέπετε ότι πάρα πολλά από τα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν στην Επιτροπή μας συνδέονται με τις διαπιστώσει που κάνετε εσεί στο δικό σα χώρο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μπερέ. Κύριε Ντεβίτ, θα, θα πρέπει να σα ευχαριστήσω και πάλι εξ ονόματο όλων των συναδέλφων για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την ζωντανή συζήτηση που προκαλέσατε. Είναι μια πολύ καλή απαρχή για την επερχόμενη συζήτηση μα με τα Εθνικά Κοινοβούλια τον Νοέμβριο. Κάθε επιτυχία και στο έργο σα στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Και εφόσον δεν έχουμε τίποτα άλλο στην ημερήσια διαταξή μας, απλώς θέλω να σας πω ότι η επόμενη μας συνεδρίαση είναι στις 11 Νοεμβρίου από τις 3 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους.